την περίοδο συνόδου για το 2010, την διακόπτω καλύτερα. Σας εύχομαι καλή και ασφαλή επιστροφή στις αιστείες σας και σε αυτούς οι οποίοι